προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη ε, στον ΟΗΕ και ιδιαίτερα στην ε, τουρκική κυβέρνηση για να ενισχυθεί η συνεργασία και να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Ζασάδα. Περνάμε στις ψηφοφορίες, δεν έχουμε και πολλές για σήμερα. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η ψηφοφορία έκθεση Μάση ε, Πιντάλγο για το Γραφείο Εναρμόνηση Εσωτερικής Αγοράς με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ο κύριος Στίβενσον. Τεχνικό πρόβλημα μάλιστα. Επόμενο θέμα. Έκθεση Λέχνερ. Τεχνικό πρόβλημα έχει και το μηχάνημα του κ. Καζίνη. Άλλος κανείς. Το ίδιο και η συνάδελφος. Και εγώ έχω πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, και ελπίζω να διευθετηθεί ο Σονούπο, γιατί κυκλοφορεί ένας τεχνικός. Μάλιστα, ας προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε το επόμενο θέμα, την έκθεση Λέχνερ, για τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρών, καθώς και των μητρών εταιριών. Με ονομαστική κλίση, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Λέχνερ. Ξέχασα προηγουμένως να συγχαρώ και τον κύριο Μάση Πιεντάλγο. Μπράβο και στους δυο σας. Επόμενη έκθεση του κυρίου Χάγκλουντ για το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Γουινέας Μπισάο για τον καθορισμό αλληλευτικών δυνατοτήτων. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτή. Συγχαρητήρια κύριε Χάγκλουντ. Επόμενο θέμα, έκθεση Nets για τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στα προγράμματα της Ένωσης. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Νέιτς. Συγχαρητήρια και στους Μαροκινούς Αλείς. Επόμενο θέμα. Ε, σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της ε, ε πρόταση του Συμβουλίου για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Το λόγο έχει ο εισηγητή ο κύριος Βοητσεχόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, οριστικοποιούμε σε μια πολύ σημαντική εργασία για ένα κανονισμό που διευκολύνει τον εμβολιασμό ε, κατά μιας πολύ σοβαρής επιζώτιας που ε, απειλεί την ε, κτηνοτροφία σε πολλές χώρες. Έχουμε καλύτερα εμβόλια, καλύτερη πρόσβαση του εμβολιασμού και θα ήθελα να σας συστήσω να τη δεχτούμε ανεπιφύλακτα γιατί αυτός ο κανονισμό είναι απαραίτητος για τους κτηνοτρόφους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν χρονοφόρα η, χρονοβόρα η διαδικασία. Επιτέλους τη διεκπεραιώνουμε. Σα ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και σα παρακαλώ να υποστηρίξετε την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Thank you. Well, as no... Μια ναι, και δεν έχουν υποβληθεί προτάσει για απόρριψη τη θέση του Συμβουλίου και δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίε, ε, εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου και ευχαριστούμε τον κύριο Βοτσεχόφσκι. Επόμενη έκθεση τη κυρία Εσάια για τεχνικέ απαιτήσει για τι μεταφορέ πίστοση και τι άμεσε χρεώσει σε ευρώ. Εσάια. Πρώτη ομάδα τροπολογιών. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την ούτω τροποποιηθεί σε πρόταση Επιτροπή. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματο. Ποιο είναι υπέρ. Α, υπάρχει μια τροπολογία, συγγνώμη. Τροπολογία 111. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Και συγχαρητήρια κυρία Σάια. Επόμενο θέμα. Έκθεση για άλλα σέντερ για τον ορισμό ενός μέλους του ελεκτικού συνεδρίου. Το κύριο μπαουντηλιο Τόμε Μουγκουρούσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σβόμποντα που εκπροσωπεί την εισηγήτρια. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Έχω μία ερώτηση προς τον εισηγητή. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε ψηφίσει την τροπολογία σχετικά με το ελεγκτικό συνέδριο. αυτός τον οποίο είχαμε ψηφίσει από πλευράς Ισπανίας είχε παρετηθεί ή αποσύρθηκε από την Ισπανική κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι έγινε. Εμείς ψηφίσαμε για ένα μέλος λοιπόν και το Συμβούλιο δεν σέβεται από ό,τι φαίνεται την ψηφοφορία μας. Διαρωτώ με τι ακριβώς γίνεται γιατί εμείς διαμαρτυρόμεθα εναντίον του Συμβουλίου γιατί αγνοεί την ψήφο κατά πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν σέβεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο. Uh, από ό,τι φαίνεται η εντολή λύγει στο τέλος του μήνα ε, των ελεγκτών. Οπότε η πρόταση του Συμβουλίου είναι από ό,τι μου λένε σωστή. Λοιπόν, The blue vote is open. μυστική ψηφοφορία. The blue vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. ...310 υπέρ, 276 κατά 87 αποχές, δεκτή η πρόταση. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Κλείσαμε με τις ψηφοφορίες.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 Right. Um, explanations of vote. ψήφου. Η κυρία Σουίντμπερν.